Πολύ καλημέρα σας, αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι. Έχω μία ανακοίνωση. Ζητήθηκε από τον κύριο Πυρίλο διαδικαστικό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Στο... Στην πόλη Πάολα. Είχαμε χθε το βράδυ μία φοβερή καταιγίδα με προβλήματα στο ηλεκτρικό δίκτυο και ένα μεγάλο αριθμό των οικογενειών που χρειάστηκε να εγκαταλείψουν τις κατοικίες τους, έκλεισαν σχολεία και στην Καλαβρία έχουμε όλο και περισσότερο ακραία μετεωρολογικά φαινόμενα. Βέβαια, κηρύξαμε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης και ελπίζουμε ότι θα ενεργοποιηθεί το Ταμείο Αλληλεγγύης για να αποζημιωθούν τα θύματα αυτής τη καταγγελίας. Θα ήθελα να εκφράσω την αλληλεγγύη μου προς τους πληγέντες πληθυσμούς και ελπίζω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να εκφράσει την αλληλεγγύη του. Φυσικά και εμείς ανησυχούμε και εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας για αυτή την θεομηνία που έπληξε την Καλαβρία. Και φυσικά σύσσωμα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αισθάνεται αλληλεγγύη με όσου υποφέρουν αυτή τη στιγμή στην πανέμορφη περιοχή τη Ιταλία και τη Ευρώπη. Το πρώτο σημείο τη ημερήσια διάταξη προβλέπει δήλωση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τι μεταρρυθμίσει που γίνονται και τι εξελίξει τη Δημοκρατία τη Μολδαβία. Εκ μέρου τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μα παρουσιάσει το θέμα ο Επίτρεπος Φίλε. Έχετε το λόγο κύριε Φίλε. Good morning, Mr. Chairman. Καλημέρα κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές. Όταν εξετάζουμε τις σχέσεις μας με τη Μολδαβία, νομίζω πως θα συμφωνήσουν όλοι πως έχουμε επιτύχει μεγάλη πρόοδο σε χρόνο ρεκόρ. Εσωτερικά όμως